Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Ανισλάφ Μπορτζάκ μου διαβίβασε ένα αίτημα υπεράσπισης το εισασυλίας του στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διοικητικής που έχει ξεκινήσει ε, ε, εναντίον του από την υπηρεσία δημόσιων μεταφορών της Ζήλαβα. Σύμφωνα με τον κανονισμό διαβίβασα το αίτημά του στη